Ladies and gentlemen, dear colleagues. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα να συνεχίσουμε την συνεδρία της Επιτροπής μας. Χαιρετίζουμε όσους είναι εδώ. Επανερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μεγκλένα Κούνεβα, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η πρέσβυρα Κούνεβα έχει αναλάβει τα καθήκοντά της εδώ και ένα χρόνο. Είχαμε διμερή συνάντηση στο Στρασβούργο στις αρχές του έτους και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους καταφέραμε να διοργανώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ καλές σχέσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά κοινέ αποστολές εκλογικών παρατηρητών, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ που είναι από τις πιο ορατές πτυχές της ε, κοινοβουλευτικής μας συνεργασίας. Άλλα σώματα της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως είναι η Επιτροπή της Βενετίας ή το Γκρέκο επίσης ε, τροφοδοτούν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στοιχεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και εδώ στην ΑΦΕΤ, στις εκθέσεις για τη διεύρυνση, την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και βεβαίως θα συνεχίσουμε το έργο μας σύντομα εδώ στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Στο Στρασβούργο λοιπόν έχει την έδρα της η κυρία Κούνεβα, θα είμαστε και εντός του μήνα στο Στρασβούργο και εμείς, ίσως είναι και αυτό μια ευκαιρία για να ξανασυνδυθούμε. Σας καλωσορίζουμε και Θέλουμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Θα σας πρότεινα να μας ε, παρουσιάσετε την κατάσταση που επικρατεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης για 10-15 λεπτά και από εκεί και πέρα θα γίνουν και κάποιες ερωταπαντήσεις. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι προνόμιό μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη σημαντική ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα να ξεκινήσω με αυτό που ξεκινήσατε κι εσείς ότι πολύ συχνά έρχεστε στο Στρασβούργο και με πολύ μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να συνεχίσουμε σε κάθε επίπεδο αυτή τη συνεργασία. Οποτεδήποτε θέλετε να με συμβουλεύεστε ή να συζητάτε μαζί μου, είτε με μένα είτε με άλλους αξιωματήχους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ξέρετε ότι έχουμε και ένα νέο εκλεγέντα γενικό γραμματέα. Ελπίζω πραγματικά να έχουμε μια επικοδομητική και γόνιμη συνεργασία. Ε, η ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι γνωστή, όπως και ο τρόπος συνεργασίας μας. Ωστόσο, για πληρότητα θα, και σαφήνεια θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα σημαντικότερα ε, στοιχεία, ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μας. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά πρέπει να εξηγούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι το ίδιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι, είναι, είναι θέμα, είναι ζήτημα αυτό. Και είναι πρόβλημα πολλές φορές, διότι είμαστε ξεχωριστοί θεσμοί, έχουμε διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεργάζεται με 47 κράτη-μέλη για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Σε ολόκληρη την Ήπειρο και πέραν αυτής υπάρχουν κάποιες βασικά θεσμικά όργανα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι το ισχυρότερο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Έχουμε την Επιτροπή της ε, Βενετίας, τον ε, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτοί είναι κάποιοι από τους θεσμούς που ε, εντάσσονται στο επίπεδο, στο πλαίσιο του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης και βεβαίως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση επίσης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσφορά νομικών μέσων υπεράσπισης των θυμάτων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλάζουμε δηλαδή πραγματικά τη ζωή όταν ακριβώς προσφέροντάς τους μέσα προσφυγής ε, και εξασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη ε, μέσω του συστήματος που του προσφέρουμε. Τα, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την συνεργασία των 28 κρατών μελών της μέσω της εναρμόνισης πολιτικών και οικονομικών κανόνων. Όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλη της Συμβουλίου τη Ευρώπη και βεβαίω συμμερίζονται τι θεμελιώδει αξίε που ε, διακρίνουν το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και στην, στην Ευρώπη και στην περιοχή της γειτονίας. Και αυτή η συνεργασία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, την, την εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο οργανώσεων και στο τέλος έχει και απότερο σκοπό την ε, δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεργασία. Μεταξύ των δύο ε, οργανώσεων η συνεργασία έχει προχωρήσει πολύ από το 1993 όταν και εγκρίθηκε το πρώτο ε, κοινό πρόγραμμα και διαδικασία που κορυφώθηκε και με την υπογραφή ενός μνημονίου αλληλοκατανόηση του 2007, όπου πραγματικά κατοχυρώνονται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη ως βασικές αρχές, καθώς και η δήλωση προθέσεων του 2014, όπου ε, πλέον καθορίζονται αναδιετία ε, οι βασικότερες προτεραιότητες της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Του χρόνου θα γίνει η επόμενη τέτοια διαδικασία. Αυτό το πλαίσιο αναφοράς που ε, αφορά την στρατηγική ε, και διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανώσεων έχει στεφτεί με επιτυχία. Το 2018 στέφθηκε από ε, μια εντατική συνεργασία, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, συναφών θεμάτων, την ανάγκη να ενισχυθεί και να προστατευτεί η δημοκρατία και να ενισχυθούν οι κανόνε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Οι δύο οργανώσει συμμεζόμαστε τι ίδιε αξίε όσον αφορά τι δεσμεύσει για μια αποτελεσματική πολυμέρεια στον κόσμο και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το δεδομένο. Πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε αυτό το πολυμερές ε, πλαίσιο στον κόσμο, ιδίως ε, για τα σημαντικότερα παγκόσμια θέματα. Η συνεργασία των δύο οργανώσεων 2018-2019 βασίζονται και στο ε, σύστημα των συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 200 στον αριθμό, που αποτελούν μια στέρεη βάση για τη συνεργασία και αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες των δύο οργανισμών. Έχουμε ε, γραφεία διασύνδεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ στις Βρυξέλλες και ξέρω ότι εδώ ο συνάδελφος ε, είναι μαζί μας στην αίθουσα και υπάρχει βεβαίως και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο όπου ε, εγώ ε, συναντώ συχνά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπου έχουμε την ευκαιρία να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Η συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης βασίζεται στον πολιτικό διάλογο, τα έργα συνεργασίας και την νομική συνεργασία. Ξεκινώντας με τον πρώτο πυλώνα, την συνεργασία σε πολιτικό, τεχνικό επίπεδο ε, γίνονται ανοιχτέ, ειλικρινές, συζητήσει, κάτι που είναι αξιονική σημασία για την συνεργασία μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επαφές μεταξύ των, μεταξύ των δικών μας αξιωματούχων, με επιτρόπους, με τον κύριο Γιούγκερ, με την ε, κυρία Μογκερίνη, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε και την ετήσια συνάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Υψηλών Αξιωματούχων, που είναι σαν σύνοδος κορυφής αν θέλετε, καθώς εκεί γίνεται ένας απολογισμός της συνεργασίας μας και εκεί καθορίζονται και συγκεκριμένε ε, καθοδιευθυντήριες γραμμές για την ε, μελλοντική συνεργασία μας. Το Συμβουλίο της Ευρώπης και το, η Κομισιόν τρέχουν μια σειρά από κοινά προγράμματα, που είναι ο δεύτερο πυλώνα τη συνεργασία μα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να είναι ειδικά για κάθε χώρα, περιφερειακά ή πολυμερή. Για την ανύψωση των προτύπων για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στι γειτονικέ χώρε. Τα κοινά προγράμματα υποστηρίζουν νομικέ και θεσμικέ μεταρρυθμίσει σε πολλού τομεί και περιλαμβάνουν διάφορε δραστηριότητε, όπω ε, εκπαιδευτικοί κύκλοι, σεμινάρια, ε, παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες σε κυβερνήσεις, όλα αυτά σε συνεργασία πάντοτε με τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών. Τα κοινά προγράμματα αποτελούν τον κυριότερο πόρο τη συγχρηματοδότηση από την πλευρά Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόθεση τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου, δικαίου στην ε, νοτιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία, τον Κάφκασο, την ε, Κεντρική Ασία και αλλού. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ενισχύει τον ορατό του και προβλέψιμο ρόλο του στα προγράμματα αυτά. Το 2018 ε, υλοποιήθηκαν 52 τέτοια κοινά προγράμματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέσω των περιφερειακών του γραφείων σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα κοινά προγράμματα μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως, σκοπό την προώθηση της ανθρώπινης δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και αποτελούν το βασικό πυρήνα και την πηγή χρηματοδότησης τεχνικής αρρωγής που παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις άλλες χώρες. Το 2018 ε, τα χρήματα των χρηματοδοτήσεων ανήλθαν σε 152,8 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθαν τα 131,4 εκατομμύρια ευρώ, ε, πάνω από 80% δηλαδή, και 23,4%, 15% δηλαδή το, της συνολικής χρηματοδότησης. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική συνδρομή από τη δική μας πλευρά. Θέλω να σας πω ε, τι, τι, ποιο είναι το πεδίο ε, ε, εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων. Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία, προγράμματα διεύρυ, διεύρυνσης. Ε, μετά την πρώτη φάση, ανάμεσα στο 2016 και το 2019, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και τα παραδοτέα του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σαφή στόχο και προσανατολισμό το 2020. Η δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο με 35 ε, εκατομμύρια ευρώ έως το 2021. Το, το επόμενο είναι η ανατολική εταιρική σχέση. Μέσω της εταιρικής αυτής σχέσης για την καλή διακυβέρνηση θα έχετε δει ίσως την συντομογραφία PGG που βρίσκεται πλέον στη φάση 2 ε, έχουμε στη διάθεσή μας 17,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019-2021 και από αυτά θα καλυφθούν κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες στην ανατολική εταιρική σχέση όσον αφορά την δικαστική μεταρρύθμιση, όπως ακριβώς αυτά καθορίζονται στην ε, στρατηγική για το 2020, όπως έχουν συμφωνηθεί και στην Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική ε, Εταιρική Σχέση. Και τέλος υπάρχει και το πρόγραμμα για την ε, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που πλέον βρίσκεται στην τρίτη φάση του, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 με χρηματοδότηση 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι προτεραιότητες εκεί είναι η δημιουργία ενός νομικού χώρου πρόθεση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντίστοιχου νομικού πλαισίου, εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, ανάπτυξη ικανοτήτων και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Και τρίτος πυλώνας, νομική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, φορέων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή είναι, αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος τρόπος που έχουμε για τη συνεργασία μας την διοργανωκή. Έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει δώσει έμφαση στον ε, λόγο, έχει δώσει ιδιαίτερο ρόλο στην ε, Γκρέκο, την ε, Επιτροπή της Βενετίας. Γκρέκο είναι η ομάδα κατά της διαφθοράς που έχει σοβαρό έργο και στην καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Συνεχίζουμε το έργο μας αυτό με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ε, και ε, έχουμε και ε, καθεστώς παρατηρητή στην Κρέκο ε, ξεχωριστά. Παρά το γεγονός ότι και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν έτσι και αλλιώς σε αυτήν την σύμβαση. Και τέλος για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι υποχρέωση κάτω, με βάση την συνθήκη της Λισαβόνας και είναι το σημαντικότερο βήμα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θα δώσω τη δυνατότητα αυτό ε, στο ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου να εκδίδει αποφάσεις και είναι γνωστό ότι πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητα αυτής της σύμβασης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ξεκίνησαν κάποιοι, ε, κάποιες συζητήσεις, επαφές που βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα φάση αυτών των συζητήσεων και ελπίζω, δεν έχουν ολοκληρωθεί και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να επανέλθω και να σας ενημερώσω με βάση τις εξελίξεις που θα έχουμε πιο συγκεκριμένε. Πάντως, ε, εργαζόμαστε πολύ καλά και στον τομέα της ε, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε νέο γενικό γραμματέα που εξελέγει πρόσφατα είναι ε, είναι μια γνωστή ε, Ευρωπαία πολιτικός, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας, η Μαρίνα Μπούριτς. Νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει μια νέα όθηση στη δουλειά μας, μια νέα ορμή, η εκλογή της δηλαδή, και ενδεχομένως να ε, ε ακουσούν και κάποιες ερωτήσεις για για την ε, Ρωσία. Ε, να σας πω και δύο λόγια γι' αυτό. Έχουμε μια συζήτηση για την διαδικασία συμπληρωματικότητας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της, του Συμβουλίου που θα ξεκαθαρίσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι δύο θεσμικοί αυτοί φορείς και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δείξουμε σε όλα τα κράτη-μέλη ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και ότι προστατεύουμε και υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση και σε κάθε περίπτωση την, τις αξίες μας. Νομίζουμε ότι η πολυμέρεια είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε τοπικά, εθνικά, περιφερειακά συμφέροντα, πάντοτε με τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τέλος νομίζω ότι ε, αυτός είναι ένας εξαιρετικός δρόμος, ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναπτύξουμε αυτά που βρίσκονται πραγματικά στον πυρήνα της ίδιας μας της ύπαρξης, να είμαστε μαζί, να συμβιώνουμε. Αυτό αυτό είναι και ε, το κέντρο του, του γνωστού πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι που έχει πραγματικά τον, ε, τον ε, άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος. Αυτό είναι και δικός μας σκοπός. Πάντοτε με διάθεση και σκοπό να μεταλαμπαδεύσουμε τις δικές μας αξίες και ε, τη δική μας αισιοδοξία και προς τα έξω και νομίζω ότι και ο δικός μου φορέας αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πραγματικά ο κατάλληλος χώρος για να ακουστεί αυτή η ευρωπαϊκή φωνή. Ευχαριστώ κυρία Κούνεβα για την παρουσίαση. Έχουμε περίπου 20-25 λεπτά στη διάθεσή μας ε, κυρίες και κύριοι για τις ρωταπαντήσεις. Να μονοστοποιήσετε αν θέλετε το λόγο. Το επόμενο σημείο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και τον πρέσβη κ. Σάτλα. Ε, τώρα όμως μιλάμε για το Συμβουλίο της Ευρώπης. Όλοι περιμένουν την 18 Σεπτεμβρίου όταν θα, ορκιστεί η καινούρια ε, γενική γραμματέα, όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα, αλλά είναι και από ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί από εσά, από εμά εδώ τη γνωρίζουμε και προσωπικά. Ε, ίσως κάποια στιγμή, και το λέω ευγενικά, αφού είστε στο Στρασβούργο και εμείς είμαστε τουλάχιστον μια φορά το μήνα στο Στρασβούργο, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πρωι, πρωινό, παραδείγματος ένα πρόγευμα συζήτηση ε, συζήτησης, έτσι ώστε ε, να μπορούμε να συζητούμε μια σειρά από Αυτή είναι η επιθυμία μου για το επόμενο έτος, η ευχή μου. Ε, και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη μα να είστε σύντομοι παρακαλώ. Η κυρία Σόφκο πρώτα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την κυρία Πρέσβη. Είμαι από την Κροατία και θα ήθελα και εγώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την πρώτη γυναίκα γενική γραμματέα και είναι και από τη χώρα μας μάλιστα, πρώην υπουργό Εξωτερικών και θα βοηθήσει ε, σε αυτό το έργο συντονισμού μεταξύ Συμβουλίου, και, Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, 80% του προπολογισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχουμε κάπως πιο ενεργά ε, για το να δούμε πώς λαμβάνονται τελικά οι αποφάσεις και πώς εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, διότι εδώ μιλάμε για στήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, τα οποία προφανώς ε, και απασχολούν πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχει και την νοτιοανατολική εταιρική σχέση. Μπορείτε να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα για την επιστροφή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις, ε, πώς προχωράει αυτή η συνεργασία και επίσης υπάρχει το θέμα της Τουρκίας που δεν σέβεται πολλές από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, ε πώς προχωράει ο διάλογος και η συνεργασία με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο και ο Σκομπίλη, ο κ. Γκάρνερ, ο κ. Λούντενοφ, ο κ. Λαγκουντίνσκι και ο κ. Μαριανή. Ε, έχω ξεχάσει κάποιον. Λοιπόν, εντάξει, αυτοί είναι οι ομιλητέ. Α ακούσουμε λοιπόν όλου του ομιλητέ για να απαντήσετε στο τέλο. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θέλετε να απαντήσετε στον καθένα ξεχωριστά, όχι, σε όλου μαζί. Λοιπόν, για τους πράσινους η Χέλα Γκουντίνσκι έχει το λόγο, ο κύριος Γκουντίνσκι, συγγνώμη, έχει το λόγο. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ, λέει ο κύριος Λαγκουντίνσκι. Για την Τουρκία θέλω να μιλήσω, έχω δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα, από το 2007 υπάρχει μια συνεργασία ε, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση στον δικαστικό τομέα με την Τουρκία υπό το φω της κατάστασης στην Τουρκία, δεν χρειάζεται τώρα να τα εξηγώ, ξέρετε τι γίνεται ιδιαίτερα στο δικαστικό τομέα, ε, πού βρίσκεται αυτή η συνεργασία, συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης, ε, είναι εφικτό να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Δεύτερο ερώτημα, πάλι για την Τουρκία. Έγιναν ε, κάποιες επισκέψεις από το 2016 και τελευταία το 2019 ε, όπου ε, έλαβα χώρο συνεντεύξεις στους πολιτικούς κρατουμένους στα πλαίσια της Επιτροπής ε, ε, κατά των, ε, της παραβίασης των δικαιωμάτων εκεί. Δεν έχουμε κανένα νέο όμως από αυτές τις συνεντεύξεις, δεν υπάρχει κάποια έκθεση. Τι συνέβη, θα δημοσιευθεί κάτι, ενημερώστε μας. Επίσης, ποια είναι η δική σας θέση για την κατάσταση με τη Ρωσία υπό το φως βέβαια του η Ρωσία επέστρεψε ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως πλήρες μέλος ε, και τα λίγα κοινωνικά δικαιώματα που παραμένουν στη Ρωσία αυτή τη στιγμή καταπατώνται την ίδια στιγμή. Ποια είναι η θέση σας λοιπόν από αυτού. Ευχαριστώ και κύριος Μαριανή έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε γνωρίζω το Συμβούλιο τη Ευρώπη, ήμουν 10 χρόνια εκεί, ε, ήμουν στην ε, πρόεδρο τη Επιτροπή Monitoring, να πω ε, δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα για το κείμενο σχετικά με την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανησυχούμε όλο και περισσότερο. Στα πλαίσια τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία, αμφισβητούμε όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα αυτών των εξαιρετικά προβληματικών τη ε, δήλωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια δήλωση που τελικά αντί να εγγυάται την ασφάλεια προσπίσει τα, ε, τα δικαιώματα των τρομοκρατών. Ε, ο Καμέλ Ντουαντί, α πούμε, τρομοκράτη, ε, δεν μπορούμε να το στείλουμε στην Αλγερία πίσω διότι το Συμβούλιο ε, ή μάλλον μια απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μα το απαγορεύει και τον στέλνουμε από μια πόλη στην άλλη. Δεν νομίζετε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει ε, αυτό, αυτή η ολίσθηση του, ε, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, τώρα, για την εκλογή των δικαστών εκεί, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχα συμμετάσχει στην εκλογή του δικαστή από τη Μακεδονία το 2016, ο οποίο δεν πληρούσε κανένα στοιχείο, κανένα, καμιά προπόθεση, κανένα προσόν. Δεν ήξερε ούτε αγγλικά ούτε γαλλικά, γαλλικά καθόλου και αγγλικά σαν ένα εξάχρονο παιδάκι και δεν γνώρισε κανένα άρθρο τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καμία απόφαση του δικαστηρίου και στην Επιτροπή μας του, δώσαμε εμείς τη σύμβαση για να δείξει μια ματιά και να πει δύο λέξεις. Αυτή η διαδικασία, η οποία είναι τελείως πολιτικοποιημένη του ορισμού των δικαστών στην, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πληρεί σήμερα ε, τι προποθέσει αποτελεσματικότητα. Επίση, εγώ χαίρομαι που επιστρέφει η Ρωσία, αλλά η Ρωσία επέτρεψε κυρίω επειδή η Τουρκία πλέον έχει κόψει ε, τη μισή συμμετοχή της. Η Ρωσία είχε αποσύρει ολόκληρη τη συμμετοχή τη Μήπω τελικά δεχτήκαμε τη Ρωσία, που εγώ χαίρομαι που στρέφει η Ρωσία, μήπω τελικά δεν δέχτηκε το Συμβούλιο τη Ευρώπη μόνο και μόνο για οικονομικού λόγου. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα για το ΕΛΚ, δεύτερο ομιλητή, ο κ. Κουμπίλιο. Uh, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρέσβη, χαίρομαι που είστε εδώ. Ήμουν στο και εγώ στο Στρασβούργο, προσπαθούσα να γίνω γενικός γραμματέα, αλλά τώρα είμαι εδώ, στι Βρυξέλλε. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι για τη Ρωσία. Είδα και εγώ ότι υπήρχε μια κρίση αξιών στο Συμβουλίο της Ευρώπης, στο παρελθόν, και αυτό είναι λυπηρό. Όταν εμεί ε, γίναμε τη δεκαετία του 90 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για μα τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Υπάρχουν εκεί υψηλά πρότυπα και για μας ήταν ένα, ε, ένα πρώτο βήμα για να γίνουμε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόσουμε αυτά τα πρότυπα και στη χώρα μας. Τώρα όμω ε, έχουμε τη Ρωσία η οποία επέστρεψε και που συμπεριφέρεται, υποτίθεται, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Είδαμε όμως τι γίνεται στη Μόσχα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και, της και τη Ρωσία. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ρωσία βελτίωσε τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία ή το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν αυτό που ε, υποτίμησε τα δικά, τα του πρότυπα. Ευχαριστώ κύριε Κουμπίλιουσο. Μίχελ Γκάλα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και πολλές δεκαετίες το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το κλαμπ της δημοκρατίας των ε, κρατών που η δημοκρατία λειτουργούσε. Και νομίζω ότι δικαίως συμμετέχει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη μεριά η είσοδος εκεί της Ρωσίας στη δεκαετία του 90 συνοδεύτηκε από πολλές ελπίδες. Τελικά όμως, τι είχαμε. Είχαμε την προσάρτηση της Κρυμαίας, την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια αυτής της επίθεσης, το 2014, όταν κάναμε ψηφίσματα εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, Βλέπουμε λοιπόν τι έχει γίνει εντωμεταξύ. Ότι χωρίς όρους δεχτήκαμε και πάλι πίσω την Ρωσία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εκπροσωπείται εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα διατηρεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Εσείς λοιπόν εκπροσωπείτε έναν θεσμό ο οποίος αναγνωρίζει βεβαίως ότι συνεχίζεται η επίθεση εκεί, αλλά διατηρεί την Ρωσία στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα μπορούσατε λοιπόν να επιμείνετε ούτω ώστε τουλάχιστον οι προσδοκίες που είχαμε εναντί της Ρωσίας αυτά που περιμένουμε από τη Ρωσία να γίνουν πέρα από λόγια και πράξει. Είστε σε θέση να επιμείνετε λοιπόν ενώπιον των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ούτως ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά που ε, έχουν υποσχεθεί. Νομίζω ότι είναι λοιπόν κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε. Να δείτε λοιπόν αν όλα αυτά που περιμέναμε μέσω όλων αυτών των ψηφισμάτων από την Ρωσία να έχουν τελικά εφαρμοστεί. Και θα ήλπιζα να είναι ο ρόλος σας, διότι μας εκπροσωπείτε και εκπροσωπείτε λοιπόν και εμάς όσον αφορά το θέμα με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιόντανοφ, ο βουλγάρος συμπατριώτης σας, κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κούνεβα, θα μιλήσω βουλγάρικα. Ξέρετε ότι γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Ήσασταν υπουργό μου. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι όταν ήμουν πρόεδρος του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου η Βουλγαρία ε, έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αν τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία επικρατούσε ένα καθεστώς που βλέπουμε σήμερα να υπάρχει στη Ρωσία, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα είχαμε γίνει δεκτή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα συνεχίσω στο ίδιο μήκο κίνηματο που μίλησαν και οι συνάδελφοί μου. Η Βουλγαρία ανησυχεί βαθύτατα για το αντιδημοκρατικό καθεστώς ε, Πούτιν. Μας ανησυχεί πάρα πολύ η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 400 χιλιόμετρα από την πόλη από την οποία κατάγομαι εγώ, τη Βάρνα. Που είναι και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο, μόνο ο εύξηνο πόντος μας χωρίζει εμά από αυτήν την τόσο επιθετική χώρα. Θεωρώ ότι η Μόσχα συνεχίζει να διώκει υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να διαλύει και να καταστέλει ειρηνικέ διαδηλώσει και διαμαρτυρίες ανθρώπων δηλαδή που θέλουν ως πολίτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες. Οι φυλακές είναι γεμάτες πολιτικούς κρατομένους και βλέπουμε να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η τραγωδία ανθρώπων όπως ο Όλεξ Εξέντσοφ και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει γίνει η ανταλλαγή κρατουμένων και ακούμε και τις τελευταίες διακηρύξεις του κυρίου Πούτιν που είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τη συμφωνία του Μίνσκ και ότι η Κρυμαία θα συνεχίσει να είναι έδαφος προσαρτημένο, κατεχόμενο και οι μόνες διαμαρτυρίες που δέχεται είναι ειρηνικές. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την, ε, της ΕΠΑ και τον Καναδά επιβάλλονται απλώς κυρώσεις ως ειρηνικό μέτρο. Εμένα το ερώτημά μου είναι τι μπορεί συγκεκριμένα να κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου, τι μπορεί να κάνουν με σκοπό να επανέλθει η Ρωσία, όσο αφηρημένο και αν ακούγεται αυτό που θα πω, να επανέλθει λοιπόν η Ρωσία στον δρόμο της προστασίας και της υπεράσπισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Γιόρντανοφ. Πολλά ακούστηκαν. Κυρία Κούνεβα, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής ε, στις περισσότερες ερωτήσεις που ακούσαμε. Γι' αυτό θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω τον όρο κοινέ ανησυχίες, αν θέλετε. Και σε αυτές τις, αυτές τις ανησυχίες τις συμμερίζομαι και εγώ προσωπικά ως ε, Ευρωπαία διπλωμάτης. Με ενδιαφέρει πολύ πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των πολιτών στην Ρωσική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα ε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία από τη δική μας πλευρά. Θέλω όμως να σας πω ποιες ήταν οι πρόσφατες εξελίξεις με τη Ρωσία για να ξέρετε και εσείς πού βρισκόμαστε. Η Ρωσία ε, εκδιώχθηκε από το ΠΕΙΣ, από την Κοινοβουλική Συνέλευση, της αφαιρέθηκαν δηλαδή τα, ε, τα δικαιώματα ψήφου της. Αλλά αυτό είναι, ένα από, είναι ένας από τους φορείς. Του στερήθηκαν λοιπόν τα δικαιώματα ψήφους, για, ψήφου για πέντε χρόνια, όμως ποτέ ποτέ οι Ρώσοι δεν στερήθηκαν το δικαίωμα να παρίστανται και να ε, έχουν δικαίωμα ψήφου στο, στην Επιτροπή των Υπουργών. Και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί είναι διαφορετικό. Θέλω να την τονίσω αυτή την κατάσταση. Ακόμη και όταν σταμάτησαν να ε, συνεισφέρουν τη συνδρομή τους, που είναι λίγο παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ κατέτος προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, παρόλα αυτά διατήρησαν τη θέση τους στην Επιτροπή Υπουργών, που έχει στρατηγική συμμαχία σύμφωνα με το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και παρά το γεγονός ότι στην ΠΕΙΣ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση δηλαδή, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, η Επιτροπή των Υπουργών συνεδριάζει κάθε βδομάδα. Η Ρωσία ποτέ δεν έφυγε από εκεί και μάλιστα ε, το έκανε και δωρεάν, ακριβώς γιατί δεν συνεισέφερε οικονομικά πλέον. Οπότε τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Η Υπουργική Επιτροπή θα μπορούσε και να εκδιώξει την ε, ε Ρωσία βεβαίως θεωρητικά, αλλά δεν υπήρχε ε, πλειοψηφία υπέρ μιας τέτοιας επιλογής ή αλλιώς να βρεθεί μια λύση ώστε και, τα, και οι δύο φορείς, η Υπουργική Επιτροπή και η ΠΕΙΣ, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, να βρουν κοινό έδαφος. Αυτό και έγινε τώρα και αυτό για το μέλλον σημαίνει ότι, και εδώ έχω και το έγγραφο έτσι λέγεται, κοινό μηχανισμό. Είναι, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση βεβαίω και πρώτη φορά είναι πρωτοφανή αυτή η κατάσταση. Πώ μπορούν αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο φορεί να συνεργαστούν και να λαμβάνουν αποφάσει, αποφάσεις οι οποίε δεν θα έρχονται σε αντίφαση μεταξύ του. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί στο μέλλον βεβαίω. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά ε, τις εξελίξεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και ο κ. Κουμπίλιου. Ε, εδώ μαζί μας. Θυμάμαι πολύ καλά ακόμη όταν παρουσιάσατε στο Συμβούλιο της Ευρώπης την, το όραμά σας για τον τρίτο πυλώνα. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές εκθέσεις, την νομική έκθεση ε, Μπουλκοβέτσης, την ε, έκθεση Νικολέτη, την ε, έκθεση Ντεσούτα που είναι και ευρωβουλεύτρια πλέον και αυτό που θέλω να πω είναι στο τέλος ότι οι βουλευτές δεν μπορείς να τους στερήσεις δικαίωμα, το δικαίωμα ψήφου στην ΠΕΙΣ που ήταν ο, μονα, ε, μοναδικός οργανισμός στον κόσμο όπου η, ε, η Ρωσία στερήθηκε τα δικαιώματα ψήφου της. Μόνο εκεί έγινε αυτό για τη Ρωσία. Και θα ήθελα να πω, υπερασπιζόμενοι βεβαίως στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Έχουμε φτάσει στο τέλος της ιστορίας. Όχι. Γιατί κάθε χρόνο ε, οι χώρες υποβάλλουν τα διαπιστευτήριά τους. Και αυτή είναι και η ισχύς που έχει η κοινοβουλευτική συνέλευση. Μπορεί να απορρίψει τα διαπιστευτήρια που υποβάλλει κάποια χώρα. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας. Στο ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Πρέπει να επαγρυπνούμε, να κάνουμε τη φωνή μας ακουστή και να μην εφησυχάσουμε. Εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου όταν καλούμε να εκφωνήσω κάποια δήλωση ή κάποιο λόγο στην Υπουργική Επιτροπή, καταδικάζοντας πάντοτε την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με προσήλωση υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και εδαφική ακαιρεότητα της κρυμαιας απο τη ρωσια η ευρωπαικη ενωση με προσηλωση υπερασπιζεται την εθνικη κυριαρχια και εδαφικη ακεραιοτητα της ουκρανιας Και σας διαβάζω από την τελευταία μου δήλωση. Συνεχίζουμε να καταδικάζουμε την προσάρτηση της Κρυμαίας και ε, εξακολουθούμε να είμαστε προσιλωμένοι στην πολιτική μας περί μη αναγνώρισης. Σε καμία περίπτωση η συμμετοχή της ε, Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν θα αποδυναμώσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της χώρας. Το Συμβούλιο ε, εξασφαλίζει την πρόσβαση Ρώσων πολιτών στο, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γι' αυτό και θέλουμε η Ρωσία να παραμείνει στη διακοινοβουλευτική συνέλευση. Πριν από την ε, κρίσιμη συνάντηση αυτή είχα πολλέ συναντήσει με μη κυβερνητικέ οργανώσει που μα έλεγαν ότι αν η Ρωσία εγκαταλείψει το Συμβούλιο τη ε, Ευρώπη, θα, τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Είστε η έσχατη λύση μα. Δεν έχουμε πουθενά κανένα άλλο καταφύγιο. Περιμένουμε λοιπόν από τη Ρωσία να εξασφαλίσει ότι οι κυρώσει τη θα είναι ε, ευθυγραμμισμένε με του κανόνε και τι αρχέ του Συμβουλίου τη Ευρώπη και να το καταδείξει αυτό με θετικό τρόπο, καθώ το Συμβούλιο τη Ευρώπη έχει δεσμευτικά πρότυπα και στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι τα πρώτα θετικά βήματα θα μπορούσαν να είναι ε, ε, η Ρωσία να επιτρέψει στην ε, Ντονέμια Άτοβιτ, την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη, να επισκεφτεί την Κρυμαία, την παρανόμω στα Κρυμαία, και με αυτό να έρθω και σε ένα άλλο θέμα και να απαντήσω λέγοντα ότι στην CPT, στην Επιτροπή για την ε, Προστασία από τα Βασανιστήρια, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε. Εγώ υποστηρίζω πλήρως το έγγραφο που, θα, που ε, θα δημοσιευθεί. Ε, ε, είμαι, υπέρ του να δημοσιευθούν τα έγγραφα αυτά, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία. Η Επιτροπή είναι υπέρ της δημοσίευσης. Ε, εμείς τα υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει όλα τα κράτη να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Εμείς την έχουμε δει την έκθεση και εγώ νομίζω ότι και εσείς ως ευρωβουλευτές δεν θα υπάρξει εμπόδιο για εσάς να έχετε πλήρη πρόσβαση στην έκθεση αυτή. Εγώ πιστεύω βεβαίως ότι πρέπει να δημοσιευτεί η έκθεση αυτή για το καλό και της κοινωνίας συνολικά. Γιατί αυτό είναι το ισχυρότερο ε, εργαλείο που έχουμε στην διάθεσή μας, στα χέρια μας, τη δημοσιότητα. Ιδίω ε, αυτήν την, ε, στην εποχή που διανύουμε, που με τόση ευκολία μπορεί κανείς να διαδώσει ένα τέτοιο έγγραφο μέσα από τα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε αυτά τα νέα που κομίζω νομίζω ότι είναι θετικά. Ανταλλαγή κρατουμένων, η Αντώνια Μιάτοβιτς είχε μια επίσκεψη, το ίδιο και η Επιτροπή για την Προστασία από τα Βασανιστήρια και η Ρωσία βεβαίως ε, κατέβαλε και τα ποσά που χρωστούσε για τα χρόνια που δεν πλήρωνε. Στην αρχή ε, σταμάτησε ε, να πληρώνει, τώρα πλέον έχει ε, εξοφλήσει πλήρως το χρέος της, κάτι που ήταν πάρα πολύ σοβαρό για εμάς και ήμασταν άτεγκτοι σε αυτήν την απέτησή μας το θεωρούσαμε, το, το παρουσιάσαμε ω απόλυτη προπόθεση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σα ξαναδεχτούμε στην κοινοβουλευτική συνέλευση αν δεν πληρώσετε τα χρέη σα. Για τα προγράμματα στην Τουρκία δικαίω ανησυχείτε. Ε, επενδύσαμε πάρα πολλά. Ε, και νομίζω ότι κάποια από τα προγράμματα στέφτηκαν τα περισσότερα προγράμματα στέφτηκαν με επιτυχία. Κάποια βεβαίως ανεστάλησαν στην υλοποίησή τους. Ε, κάποια διέρχονται μια σοβαρή ε, αναθεώρηση από κοινού γίνεται αυτή η αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε καμία περίπτωση δεν το θεωρούμε ε, το θέμα αυτό ε, δευτερεύουσα σημασία. Εγώ όποτε έχω την ευκαιρία, όταν δεν έχω την υποστήριξη όλων των κρατών ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνω μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια τοπική δήλωση, όταν, και αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές, όταν τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανιζόμαστε με μια φωνή. Και πρέπει να δείτε πόσο περήφανοι είμαστε όταν υπερασπιζόμαστε τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα είτε στην Τουρκία είτε στην ε, Ρωσία. Θα αναθεωρήσουμε λοιπόν τα προγράμματα αυτά, θα δούμε πώς προχώρησαν στην υλοποίησή τους και από πολύ στενά θα παρακολουθούμε την κατάσταση από εδώ και στο εξής. So, uh, Mariani, uh, Κύριε Μαριανή, θα σας απαντήσω για το ερώτημά σας. Νομίζω ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντιμετωπίζει βεβαίως νέες προκλήσεις, όμως κάτι για το οποίο πρέπει να είστε σίγουρος είναι ότι εφαρμόζει την νομοθεσία. Δεν εφευρίσκει η νομοθεσία, την εφαρμόζει. Την νομοθεσία και τη συμβάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν, έχετε, αν είχαμε άλλο δίκαιο, ε, εμπράγματο δίκαιο, θα είχαμε και άλλα, άλλα, άλλους δικαστές άλλες, ε, άλλες αποφάσεις. Μην αμφισβητείτε την ε, ποιότητα των δικαστών. Ε, υπάρχουν τρεις δικαστές από κάθε χώρα αυτή τη στιγμή. Και το pace είναι αυτό που αποφασίζει. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το pace να συμμετέχει στη διαδικασία. 28 δικαστές δεν έχουν εκλεγεί με την, ψηφο, με την ψήφο των, ε, της ε, Ρωσίας. Αλλά δεν νομίζω αυτό να είναι θέμα. Η εφαρμογή είναι θέμα που επανεξετάζεται κάθε χρόνο και είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία όταν εξετάζουμε τι γίνεται ε, με τα διάφορα εποπτικά όργανα, την, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αλήθεια πάντω ότι ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, μάλλον η δουλειά του, της, του Δικαστηρίου είναι πολύ, είναι πολύ, έχουν μεγάλο φόρτο εργασία. Ε, οπότε μπαίνει ένα θέμα του πώ οι δικαστέ ε, συμμετέχουν για την τελική απόφαση. Είναι πάντως είναι ένα εξάρτητο όργανο, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομά του. Ε, πάντως ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. θα παρακολουθήσουμε θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό και θα επανέλθουμε. Ε, ευχαριστώ κυρία Κούνεβα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Επίσης, να νιώσατε καλά που επιστρέψατε εδώ, στο Κοινοβούλιο. Η κυρία Κούνεβα ήταν και η πρώτη ε, βουλγάρα επίτροπος, έτσι. Ε, ήσασταν συχνά εδώ. Ναι, εμένα πάντα μου αρέσει να έρχομαι εδώ στη συνεδρία της Επιτροπής Τη επιτροπή σα, ε, κάντε μα τη χάρη. Όταν είστε στο Στρασβούργο, ενημερώστε μας ε, και να κάνουμε περισσότερες κοινέ συζητήσει. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο επόμενο χρονικό διάστημα και καλή τύχη ε, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. And all I can say is and uh, good luck. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ και καλή τύχη. Το επόμενο στήμα θα εξεταστεί για κλεισμένο των θυρών, οπότε όσοι πρέπει να φύγουν από την αίθουσα να φύγουν τώρα.